μας οδηγήσουν σε αυτή ε, τη λύση. Χρειάζεται και όραμα οικονομικό και μετά τους απαραίτητους πόρους να βρούμε για να το υλοποιήσουμε. Τώρα έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να το ε, κατευθύνουμε, να το στρίψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ράντζελ, για 1,5 λεπτό επίσης. Πρόεδρε,